Τώρα τελευταίο έκθεση του κύριου Πρέντα, φόρουμ, τέταρτο φόρουμ υψηλού επίπεδου για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας. Τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Το τέταρτο φόρουμ υψηλού επίπεδου για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας που θα γίνει στον Πουσάν τον Νοέμβριο δίνει την δυνατότητα να εμβαθύνουμε και να επαναδιατυπώσουμε ούτως ώστε η βοήθεια να λειτουργήσει καλύτερα και να προωθήσουμε την ανάπτυξη. Οι προσδοκίες είναι σημαντικές και ελπίζουμε ότι η συνεδρίαση θα δώσει περισσότερες φιλοδοξίες για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις εν ώψη του 2015. Για να πετύχει το φόρουμ πρέπει να αντιμετωπίσουμε πολλές προκλήσεις. Πρώτον η εφαρμογή μετά από, τις, από το θέμα της, απο, του απολογισμού των, της ατζέντα του Παρισιού ε, είδαμε ότι οι καλές πρακτικές πήγανε καλά βέβαια ε, βλέπουμε ότι οι καλές πρακτικές έχουν προχωρήσει αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις ε, δεν εφαρμόζονται σωστά. Έχουμε ένα πρόβλημα με τον κώδικα συμπεριφοράς και τον καταμερισμό εργασιών. Έτσι κέρδισε η Ευρώπη 6 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Πρόκειται για μια τεράστια όμως ευκαιρία που έχασε η ανάπτυξη. Η πρώτη όμως πρόκληση είναι καθαρά πολιτική, στον που σαν χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή leadership, χρειαζόμαστε δεσμεύσεις για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο στη θεματική της αναπτυξιακής βοήθειας. Χρειάζεται και η πρόκληση της προσαρμογής. Ο σκληρός ε, πυρήνας με τις πέντε αρχές ε, για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας δεν θα πρέπει να ξεχαστεί. Πρέπει να αποτελέσει τη βάση για να οικοδομήσουμε. Αλλά χρειάζεται να βρεθούν και νέοι δότες, νέοι δωρητές, εμπλοκή των ιδιωτών ε, συνεργασία μεταξύ νότου-νότου για να μπορέσουμε να έχουμε πιο αποτελεσματική βοήθεια. Χρειάζεται λοιπόν στον Μπουσάν να αναπτύξουμε σημαντικά και απαρτεναριά για την συνεργασία. Η έκθεση μου διαπιστώνει τους τομείς όπου θα πρέπει να γίνουν περισσότερες προσπάθειες για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας δημοκρατία, συνεργασία των δικιούχων, συντονισμός των δωρητών, ε, κατανομή και προβλεψιμότητα της βοήθειας. Υπάρχει μια σύγκληση απόψεων με την Κομισιόν η οποία στις 7 Σεπτεμβρίου πρότεινε να έχουμε μια κοινή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη συνεδρίαση του Μπουσάν και βασιζόμενη στα ίδια στοιχεία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας από το Φόρουμ του Παρισιού και αυτό και μέσα από τη συνεδρίαση της Άκρα για να μπορέσουν να προχωρήσουν με συγκεκριμένες δεσμεύσεις πάνω από το 50% της ε, αναπτυξιακής βοήθειας ε, δίνεται από την Ένωση και η συνθήκη της Λισαβόνας έχει δώσει προτεραιότητα στην καταπολέμηση της φτώχειας. Περιμένουμε ενισχυμένα αποτελέσματα λοιπόν στον τομέα της ανάπτυξης. Λαμβάνοντα υπόψη τώρα τι έχει γίνει στο παρελθόν πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να έχουμε μία φιλόδοξη σχέση στο, ε, θέση στο Πουφσάν. Το Συμβούλιο θα πρέπει τώρα να εγκρίνει για το τέταρτο φόρουμ μια ευρωπαϊκή κοινή θέση. Η έκθεσή μου αποτελεί μια καλή βάση για να μπορέσουμε να ευθυγραμμίσουμε τα κράτη-μέλη γύρω από αυτές τις θέσεις για τις μελλοντικέ δράσεις, για την αποτελεσματικότητα στη βοήθεια. Πρέπει να μπορέσουμε να βοηθήσουμε με μια νέα συνεργασία, με ένα νέο παρτεναριά για την υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων και να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο συντονισμένη δράση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Ζαμπόρσκα. Grazie, signora Presidente. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, στην προσπάθεια κατά πολέμησης της φτώχειας που συνεχίζεται και που συνεχίζεται και η προσπάθεια και η φτώχεια, θεωρούμε ότι η ανθρωπότητα έχουμε τα φόρα των Παρισίων της Άκρα και τα κριτήρια της Άκρας και τα κριτήρια των Παρισίων πρέπει να διασφαλίζουν ότι η βοήθεια που θα χορηγείται θα είναι αποτελεσματική. Το θέμα είναι να, να εξετάσουμε και να δούμε κατά πόσο βοηθήσαμε χρησιμοποιώντας αυτά τα κριτήρια. Στο Μπουσάν αυτό που έχουμε είναι η δυνατότητα να επισκοπήσουμε τον περίγυρο και να δούμε πού βρισκόμαστε. Δεν πρέπει όμως να απεμπολίσουμε τον κυριότερο στόχο. Αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια αποτελεσματικά, πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να αυτοβοηθηθούν. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Ευχαριστώ. La Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον συνάδελφο Πρέδα για την έκθεση είναι πολύ σημαντική. Για την έκθεση του Μπουσάν, για τις συνεδρίες του Μπουσάν, εμείς θα πρέπει να είμαστε πολύ φιλόδοξοι για την αναπτυξιακή βοήθεια. Πρέπει να ενισχύσουμε τη διαφάνεια. Πρέπει να βοηθήσουμε στον συντονισμό και επαναλαμβάνω και την ανάγκη να αποκεντρώσουμε τις ε, διαδικασίες ε, στις χώρες ε, αποδέκτες της βοήθειας. Η εμπλοκή των τοπικών παραγόντων είναι σημαντική αν θέλουμε αποτελεσματικότητα στη βοήθεια. Έχουμε ένα σχέδιο της Health Investment Network η οποία έχει επενδύσει στις ικανότητες των διεθνών δικτύων και βοήθησε να μειωθεί κατά 50% την αθνησιμότητα των βρεφών στην Τανζανία τα τελευταία 9 χρόνια. Χρειάζεται ένα κώδικα, βέβαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατανομή εργασίας στην αναπτυξιακή πολιτική. Κορτές Λάστρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαριστώ τον κύριο Πρέδα για την έκθεσή του. Επιβεβαιώνει ότι ο αγώνας ε, για την ανάπτυξη, για την αναπτυξιακή πολιτική βοηθάει στην καταπολέμηση της φτώχειας. Θα πρέπει λοιπόν η αναπτυξιακή βοήθεια να παραμείνει προτεραιότητα. Στο Βουσάν δεν θα, είναι η μόνη στιγμή για να μπορέσουμε να ορίσουμε ε, μερικά σημεία πρόωθησης. Θα πρόκειται για σταυρική στιγμή με νέους μηχανισμούς παρακολούθησης ε, για την καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων, για αναζήτηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης όπως για παράδειγμα της ε, φορολόγησης των, χρηστών χρηματοπιστωτικών ανταλλαγών. Ένα θέμα ουσιαστικό, ε, θέμα για την Ισπανία θα είναι η ισότητα των φύλων. Πρόκειται ως κάτι το παράβατο για μας, ε, για την ισότητα των γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο της βοήθειας. Παρακαλώ να ενισχυθεί και η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών σε στον έλεγχο και στην αποτελεσματικότητα της βοήθειας. Ο Επίτροπος Πρόεδρε, αξιότιμοι Νομίζω θα αρχίσω ευχαριστώντα τον κύριο Χουάν Πρέντε για την εξαιρετική έκθεση του. Δεν υπάρχει μεγάλη προσέλευση εδώ σήμερα, δεν ακούγονται πολλέ απόψει. Παρόλα αυτά, υπάρχει σύγκληση απόψεων ανάμεσα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό το θέμα. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να προετοιμαζόμαστε βέβαια για τη διάσκεψη των Μπουσάν. Καλωσορίζω πρώτα απ' όλα το ότι Τρει τρεις βουλευτές θα μετάσχουν στην ε, αντιπροσωπή τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό θα ε, ενισχύσει το κλίμα και τη Ένωση ταυτόχρονα. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε κάποιε συγκεκριμένε ε, προκλήσει. Πρώτον, το η δήλωση του Παρισιού και το θερματολόγιο της Άκυρας σχετικά με τα όσα έχουμε καταφέρει και όπως είπε ο εισηγητής, Ε, ως δωρητές ε, δεν έχουμε καταλήξει στους δείκτες ε, που χρειαζόμαστε. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ερμηνεύσουμε τη δήλωση του Παρισιού με τρόπο ώστε να έχουμε καλύτερα ηχέγγυα για αξιόπιστα αναπτυξιακά προγράμματα για να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα της εξωτερικής βοήθειας. Όπως είπε και η αξιότιμη κυρία Ζαμπόσκα θα πρέπει να μάθουμε σε κάποιον να ψαρεύει, όχι να του δίνουμε το ψάρι. Και νομίζω ότι έτσι θα καταφέρουμε να ε, ε, επιτύχουμε τους στόχους της χιλιετίας. Ε, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε, αλλά θα βρούμε να βρούμε ένα τρόπο ώστε τα επόμενα χρόνια να επιτύχουμε με αυτούς τους δείκτες και να επιτύχει όλη η διαδικασία, διότι είναι ε, κέρια σημασία. Επίση, νέοι ναι, δωρήτε. Έχει αλλάξει το τοπίο και αν το δω από τη δική μου οπτική γωνία, επειδή είμαι για τα αναπτυξιακά ζητήματα, η Κίνα, η Ινδία και άλλε χώρε που προσφέρουν αναπτυξιακή βοήθεια δεν συμβαδίζουν με τους παραδοσιακούς εισαγωγικά δωρήτες ως προς την αποτελεσματικότητα της βοήθειας. Ε, προσπαθούμε βέβαια να δούμε τι κάνουν οι εταίροι μας, διότι ε, για να έχουμε αποτελεσματικότητα στη βοήθεια θα πρέπει όλοι να ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία, ίσως όχι με τον ίδιο ρυθμό, αλλά κυρίως με διαφάνεια, διότι η έλλειψη διαφάνειας ε, θα μπορεί να οδηγήσει σε μία επαρκή στήριξη μιας χώρας κατά την ε, καταπολέμηση της ευτόχειας. Πρέπει να εμπλακούν και οι νέοι δωρητές λοιπόν στη διαδικασία. Αυτό που έχει κέρια σημασία είναι η αύξηση της διαφάνειας. Ε, στην εποχή της ε, οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ρωτούν όλοι τι αποτελέσματα είχατε με αυτή την αναπτυξιακή βοήθεια που δίνετε. Με πλήρη διαφάνεια πρέπει να καταδείξουμε πώς χρησιμοποιούνται τα μέσα που εμείς προσφέρουμε. Εγώ μπορώ να καθησυχάσω το Κοινοβούλιο ότι δεν σημειώθηκε κατασπατάληση χρημάτων, εκατομμύρια ε, χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν, ε, γλίτωσαν από τη φτώχεια, μπόρεσαν παιδιά να πάνε στο σχολείο, αντιμέτωψαν κάποιοι χείριστες συνδίκες ε, διαβίωσης χάρη σε αυτά τα χρήματα φυσικά. Θα πρέπει να επιδιώξουμε ακόμη μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τη χρήση της αναπτυξιακής βοήθειας. Θα πρέπει από πλευράς μας να αναλάβουμε κάποιες δεσμεύσεις από πλευράς Ένωσης. πριν τον Μπουσάν, δύο πράγματα θέλουμε να επιτύχουμε διαφάνεια και εγγύηση ότι όλα τα... Υπάρχει, επικρατεί πλήρης διαφάνεια για το σύνολο των κονδυλίων που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Αναπτυξιακή Βοήθεια και δεύτερον το κοινό πρόγραμμα όλων των δωρητών. Επιτόπου θα υπάρξει σημαντικός συντονισμός, αλλά... ξέρετε ποια είναι η αδυναμία του συντονισμού. Μπορεί να το ξέρετε, αλλά μην να μπορείτε να αλλάξετε ε, μια κατάσταση. Και μπορεί κάποιοι να μην μπορούν να εκφύγουν από το εθνικό αναπτυξιακό του πρόγραμμα. Οπότε ο συντονισμό δεν επαρκεί. Γι' αυτό χρειαζόμαστε περισσότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καταλήξαμε σε αυτούς τους δείκτε. Ωραία, τώρα όμως ήρθε η ώρα να είμαστε και πιο φιλόδοξοι. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο Δηλαδή, μόνο παρακολουθώντας τα εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα θα έχουμε ε, την απαιτούμενη συνεργασία και θα εξοικονομήσουμε 5 έως 6 δις ευρώ, όπως μας είπε ε, και ο εισηγητής στην έκθεσή του. Με καλύτερη χρήση θα έχουμε ε, περισσότερα κονδύλια για την αναπτυξιακή βοήθεια χωρίς να επιβαρύνεται κανείς. Θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η διάσκεψη του Μπουσάν, πολύ θα διαφέρει από την περσινή διάσκεψη στην Κωνσταντινούπολη για τους στόχους της χιλιετίας ε, και θα είναι μεγάλη πρόκληση να συμμετάσχουν και οι αναπτυσσόμενες χώρες, οι νέοι δωρητές δηλαδή, αλλά ε, προβλέπεται επιτυχία, είναι βασική πρωτοβουλία προτού εκπνεύσει το 2015 η προθεσμία για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας. Σας ευχαριστούμε για την έκθεσή σας. Νομίζω ότι ε, όπως και στην Άγκυρα θα έχει ηγετική θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση χάρη στις προσπάθειες όλων μας. Ε, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ Επίτροπε. Ολοκληρώθηκε συζήτηση θα ψηφίσουμε αύριο στο 12.30. Θα συνεχίσουμε την Ολομέλη αύριο, 25 Οκτωβρίου, 9 με 14.